για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ε, ασφάλειας για την κατάσταση στην Ερυθρέα. Εξ της Αντιπρόεδρου της Κομισιόν και υπά της εκπροσώπου θα δώσω τον λόγο στην Υπουργό κυρία Χένις Λάσερτ. Έχετε το λόγο κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έντιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι πράγματι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψει σε σχέση με την κατάσταση στην Ερυθρέα. Αυτή η μικρή χώρα στο κέρα της Αφρικής <clears throat> εξακολουθεί να βρίσκεται στην πρώτη σελίδα των εφημερίδων γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι φεύγουν κάθε μήνα από τη χώρα αυτή. Πολλοί από αυτούς έρχονται στην Ευρώπη ζητώντας μια καλύτερη ζωή χωρίς πολιτική καταστολή και καταπίεση και καλύτερες ευκαιρίες για απασχόληση. Και παρόλα αυτά εμείς ανησυχούμε τα μάλα με τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο σεβασμός για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι βασική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εξωτερικής πολιτικής της. Και πράγματι είναι τμήμα του πολιτικού μας διαλόγου με κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο και αυτό περιλαμβάνει και τις αρχές της Ερυθρέας. <clears throat> Μέσω του διαλόγου αυτού, αλλά και με δημόσιο τρόπο εμείς εγείρουμε τις ε, ανησυχίες μας για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ερυθρέα και τονίζουμε την ανάγκη η Ερυθρέα να σεβαστεί τα βασικά δημοκρατικά δικαιώματα. Έχουμε ζητήσει να υπάρξουν συγκεκριμένες χειρονομίες όπως η απελευθέρωση κρατουμένων οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση σε κανένα εδώ και πολλά χρόνια, μεταξύ των οποίων ένα Ολλανδό πολίτη, ο κ. Ντάβι Σίσα. Θα συνεχίσουμε λοιπόν τι προσπάθειέ μα σε όλε τι ευκαιρίε να θίγουμε τα θέματα αυτά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίση θίγει ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ερυθρέα σε διεθνεί χώρου και φόρα, ιδίω στι συνεδριάσει του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ. Κάνουμε έκκληση στην Ερυθρέα να συνεργαστεί με την ε, Επιτροπή Έρευνας των Ηνωμένων Εθνών και τον Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών και να τους δώσουν πρόσβαση στη χώρα αυτή. Πιστεύουμε λοιπόν ότι μια πολιτική επαφή με τη χώρα αυτή είναι η καλύτερη επιλογή με την, για την Ευρωπαϊκή Ένωση για μια σειρά λόγων. Πρώτον, γιατί η πολιτική επαφή και ο διάλογος δίνει τη δυνατότητα να πιέσουμε για πραγματική πρόοδο και βελτίωση και μας δίνει τη δυνατότητα να επιμείνουμε για τη σημασία του να γίνονται σεβαστοί οι διεθνείς κανόνες για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η απομόνωση μιας χώρας δεν βοηθάει σε τέτοιες περιπτώσεις. Ένας δεύτερος λόγος για τον οποίο θεωρούμε ότι μια κριτική στάση εναντί της χώρας αυτής είναι ε, χρήσιμη είναι και η ένδια στη χώρα αυτή. Ανεξάρτητα από το πολιτικό καθεστώς η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δεσμευμένη να φέρει σχέδια ανάπτυξης και να βοηθήσει την ανάπτυξη στη χώρα αυτή. Πρέπει να γίνουν πολλά για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί η μεγάλη πίεση που νιώθει ο πληθυσμό τη Ερυθρέα. Οι πολίτε τη Ερυθρέα αντιμετωπίζουν μια προβληματική κατάσταση σε τροφιμικό επίπεδο και έλλειψη οικονομικών ευκαιριών. Η απόγνωσή του οδηγεί σε μια συνεχή κίνηση ανθρώπων, ιδίω νέων ανθρώπων, που προσπαθούν να φύγουν από τη χώρα τους και ακολουθούν ένα επικίνδυνο δρόμο προς την Ευρώπη και είναι εύκολη λία για τους διακίνητες. Γι' αυτό η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στο 11ο Ταμείο Ανάπτυξης θα υποστηρίξουν τις κοινωνικές ε, μεταρρυθμίσεις <clears throat> στην ε, Ερυθρέα. Υποστηρίζουν ασφάλεια σε προμήθεια ενέργειας και την οικονομική διακυβέρνηση και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Επίσης, η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης βοηθάει να υπάρξει μια πρόοδο στα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ερυθρέα. Και υπάρχει και ένα τρίτο στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Η χώρα αυτή έχει μια σταθερική θέση στο κέρα τη Αφρική, είναι γειτονική τη Αιθιοπία, του Τζιμπουτή και του Σουδάν και έχει πρόσβαση στην Ερυθρά θάλασσα και μέσω αυτή στην Αραβική Χερσόνησο. Μια σταθερή Ερυθρέα και η ελληνική Ερυθρέα που σέβεται του γειτονέ τη μπορεί να έχει ένα θετικό αντίκτυπο στη συνολική κατάσταση στην περιοχή αυτή η σύγκρουση στην Ιεμένη, οι εντάσεις στον αραβικό κόσμο, η αλλαγή των συνθήκων έχουν επιπτώσεις και στο κέρας της Αφρικής και επομένως η δική μας παρουσία θα πρέπει να βοηθήσει να ξεπεραστούν αυτές οι εντάσεις. Μια πολιτική απομόνωση δεν έχει βοηθήσει καθόλου. Η άμεση βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να βοηθήσει τις συνήκες διαβίωσης των ανθρώπων στην Ερυθρέα αποτρέπουν την πορεία αυτών προς την ζωσπαστικοποίηση και την εξτρεμιστική δράση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θέλω να βοηθήσουμε την Ερυθρέα για να συμβάλλουμε και στην περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα. Θα ήθελα να κλείσω αναφερόμενοι στο θέμα της μετανάστευσης και του ασύλου. Το Συμβούλιο αναφέρθηκε στους ε, ετούντε άσυλο από την Ερυθρέα και είπε ότι αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Είναι μία από τις μεγαλύτερες χώρες προέλευσης ετούντων άσυλο και γενικά αναγνωρίζεται σε πολύ υψηλό ε, ποσοστό η ανάγκη διεθνούς προστασίας αυτών των ατόμων. Αλλά η Ερυθρέα είναι και ενεργός εταίρος στη διαδικασία του κόνσουλ η οποία αντιμετωπίζει θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και θέματα διαχείρισης συνόρων και μετανάστευσης. Με την συζήτηση και την βελτίωση των ανθρώπων στην Ερυθρέα η παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να αντιμετωπίσει κάποιους από τους παράγοντες που εξωθούν τους Ερυθρέους σε μετανάστευση. Είναι λοιπόν ένα τμήμα της απάντησής μας στην κρίση της μετανάστευσης. Να σας πω ότι σαφώς ότι εμείς θέλουμε να σταθούμε δίπλα στην Ερυθρέα για το καλό του λαού της. Πράγματι μια κριτική <clears throat> στάση είναι και προς το δικό μας συμφέρον. Είναι ο μόνος τρόπος να προσπαθήσουμε να πιέσουμε τη χώρα αυτή να κινηθεί προ τη σωστή κατεύθυνση. Αυτό αφορά και την Ερυθρέα και άλλε χώρε. Η κριτική αντιμετώπιση επί τη βάση τη κατανόηση τη δυναμική και των προκλήσεων ενώπιών μα είναι ένα πραγματιστικό τρόπο για να μπορέσουμε να προωθήσουμε τη θετική αλλαγή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Σα ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Περνάμε στου εκπροσώπου των πολιτικών ομάδων εξ ονόματο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο. Ο κύριος Ντάβορ Ιβο Στίε. Για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, πέρυσι κάναμε μια συζήτηση για την Ερυθρέα, εδώ πέρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι περισσότερες πολιτικές ομάδες είχαν πει τότε ότι είχαν μια αρκετά σκεπτικιστική στάση απέναντι στην ιδέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δώσει την απτυξιακή βοήθεια προς την Ερυθρέα. Και είχαμε πει ότι εφόσον συνέβαινε κάτι τέτοιο, τότε θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε ζητήματα όπως σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και χρηστή διακυβέρνηση. Αυτό το οποίο βλέπουμε όμως είναι ότι παραβιάζονται συνεχώς τα ανθρώπινα δικαιώματα από το δικτατορικό καθεστώς ερυθρέα, Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τόσοι πολλοί άνθρωποι έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επικεντρώνεται κυρίως σε επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα. Και ένα πολύ μικρό τμήμα του προγράμματος αυτού έχει να κάνει με άλλου τομεί. Άρα δεν ανταποκρίνεται στα συμπεράσματα στα οποία είχαμε καταλήξει εμεί εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμεί είχαμε πει τότε ότι δεν θα έπρεπε να εγκριθεί από την Επιτροπή Ανάπτυξη το πρόγραμμα αυτό. Παρ' όλα αυτά όμω εγκρίθηκε από την Επιτροπή του EDF, από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης. Εμείς το δικό μας ψήφισμα λέμε αναφερόμενοι στην Διοργανική Συμφωνία ότι θα πρέπει τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να, να παρακολουθούν καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η Επιτροπή αυτή. Το λόγο έχει ο κύριος Νόζερ εξ ονόματος των Σοσιαλιστών. Ευχαριστώ κυρία Αντιπρόεδρε, κυρία Υπουργέ. Το θέμα τη Ερυθρέα έχει αναφερθεί σε ένα ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γιατί η κατάσταση των ανθρώπινων δικαιωμάτων στη χώρα αυτή είναι ολέθρια. Αρκεί να σα υπενθυμίσω αυτά τα οποία λέει η έκθεση της Amnesty International. Έχουμε χιλιάδε πολιτικών κρατουμένων των οποίων οι οικοί και οι οικογένειε του δεν παίρνουν καμιά πληροφορία για την κατάστασή του στις φυλακέ και για την κατάσταση των συγγενών και φίλων τους. Πιστεύω ότι θα πρέπει να τονίσουμε το γεγονός ότι η Ερθρέα συνεχώς με διάφορους ε, λόγους κηρύττει την κατάσταση εκτάκτης ανάγκης. Λένε ότι υπάρχουν προβλήματα με την Αιθιοπία και επομένως είμαστε σε μόνιμη κατάσταση εμπόλεμη. Έχουν 5 εκατομμύρια άτομα <coughs> κατοίκους από τους οποίους φεύγουν χιλιάδες κάθε μήνα προς την Ευρώπη. Η Ευρώπη προσπαθεί να επηρεάσει το θέμα αυτό με τα σχέδια της αυτά, αλλά δεν αρκεί να πούμε ότι είναι δύσκολη η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα πρέπει να ζητήσουμε πολύ περισσότερα από την Ερυθρέα. Θέλουμε ως Κοινοβούλιο να υπάρξουν πιο στεναρές αποφάσεις από την πλευρά του Συμβουλίου και της Κομισιόν και να συμμετάσχει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν βοηθάει αυτή η παρουσίαση από την Κομισιόν και το Συμβούλιο για την κατάσταση της Ερυθρέας. Ευχαριστώ. Από την ομάδα ECR έχει το λόγο ο κύριος Ντέμες Μάκια. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Υπουργέ, είναι απαραίτητο να βελτιώσουμε την κατάσταση του πληθυσμού στην Ερυθρέα. Αλλά όπως γνωρίζετε η απόφαση να να αναθεωρήσουμε το πακέτο βοήθεια στην Ερυθρέα νομίζω ότι είναι μεγάλο σφάλμα κρίσης ε, και είναι κατά της γνώμης του Κοινοβουλίου. Η Κομισιόν αποδίδει την έξοδο του πληθυσμού στην κρίση την οικονομική. Είναι σφάλμα διότι ε, δεν αναγνωρίζει ε, ότι το πραγματικό πλήγμα είναι η ολοκληρωτική διακυβέρνηση από τον πρόεδρο Αφεουέρκη. Ε, πρόκειται για μια φυλακή χώρα, συνέχεια έχουμε συνοπτικές εκτελέσεις, δεν υπάρχει ελευθερία του συνέρχεστε, του, του, του, της λατρείας ε, υπάρχει στρατιωτική θητεία επαόριστον. Τα παιδιά στρατολογούνται από τη μικρή τους ηλικία και δεν παρακολουθούν ε, τα μαθήματα της εκπαίδευσης. Έτσι εξηγείται η μεγάλη εισρωή προσφύγων στην Ευρώπη. Δεν νομίζω ότι οι αρχές θέλουν να βελτιώσουν την τύχη του πληθυσμού. Αν λάβουν περισσότερα χρήματα, απλώς θα μπορέσουν να ε, συνεχίσουν την καταπιεστική και δικτατορική τους πρακτική. Ο πληθυσμός δεν επωφελείται από τα χρήματά μας αν δεν υπάρχει στόχος αναπτυξιακός και αν δεν τηρούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα και το πράγμα πάει ακόμα πιο μακριά ακόμα και βρίσκοντας μια στέγη καλύτερη στην Ευρώπη είναι ψευδέσθηση για τον πληθυσμό διότι οι κατάσκοποι του καθεστώτος τους διώκουν ακόμα και στις ευρωπαϊκές χώρες και πρέπει να πληρώσουν φόρο επί του εισοδήματος και εδώ και χρόνια τα μέσα ενημέρωση αναφέρουν αυτές τις πρακτικές. Τα Ηνωμένα Έθνη άρχισαν μια έρευνα αλλά η Κομισιό παραμένει σιωπηλή θέλουμε πραγματικά να βοηθήσουμε αυτό το καθεστώς. Όχι. Ε, η στιγμή του θάρρους έχει έρθει. Ευχαριστώ εξ ονόματος άλλης ομάδας. Μπερτσέρα Μπαστερετσέα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βλέπουμε την ε, συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας όπου παρουσιάστηκε από την Κομισιόν και το Συμβούλιο. Αυτό είναι κάτι το επονίδιστο γιατί θεωρεί ότι με τον τρόπο αυτό μπορεί να λύσει τη διαχείριση των ε, μεταναστευτικών ρευμάτων. Το Κοινοβούλιο μας έχει τονίσει κατά, κατά επανάληψη ότι δεν μπορούμε με τέτοια βραχυπρόθεσμα και κοντόφθαλμα σχέδια να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της μετανάστευσης και του ασύλου. Και εδώ στην περίπτωση της Ερυθρέας συζητούμε την κατάσταση των, ε, της χώρας αυτής την οποία τα τελευταία χρόνια έχει δώσει εκατομμύρια επί εκατομμυρίων η Ευρωπαϊκή Ένωση για να μείνουν ε, οι πολίτε τη χώρα αυτή εκεί και να μην φύγουν. Αλλά εμεί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο χωρί να εξασφαλίσουμε ότι αυτά θα καταλήξουν στις τσέπε μια κυβέρνηση η οποία καταστέλει συστηματικά το λαό της όπως πολύ λίγες χώρε στον κόσμο. Η Επιτροπή Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην οποία είμαι μέλος, τόνισε τον προηγούμενο Νοέμβριο προς την Κομισιόν και την Υπηρεσία Εξωτερική Δράση ότι δεν πρέπει να εγκριθεί το ενδεικτικό ε, πρόγραμμα για την Ερυθρέα θα πρέπει εμείς να τονίσουμε τη θέση μας που είναι και η θέση των πολιτών που εμείς εκπροσωπούμε. Αλλά αγνοήθηκε η απόψή μας. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτά τα χρήματα για να καταστήλει ακόμα περισσότερο η Ερυθρέα μέσω του στρατού της στον πληθυσμό. Όλες οι δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Ερυθρέα είναι μονάχα να περιορίσει την στρατιωτική θητεία σε 18 μόνο μήνε. Αλλά μετά η κυβέρνηση τη Ερυθρέα είπε ότι δεν έχει καμία τέτοια πρόθεση. Μήπω θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει κάτι για να εξασφαλίσει ότι τα χρήματα των φορολογούμενων δεν καταλήγουν στα χέρια μια από τι χειρότερε δικτατορίε του κόσμου. Εμεί θα πρέπει να βοηθήσουμε να λυθούν τα προβλήματα των χωρών αυτών που είναι φτωχές και δεν θα πρέπει να σπαταλάμε έτσι, τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να διατηρήσουμε την απαραίτητη αιρεσιμότητα και τον απαιτούμενο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει και ο πρόεδρος. Από την ομάδα GUE NGL, η κυρία Μαρή Κριστίν Βέζια για δύο λεπτά. Όχι, ένα λεπτό λέει ο Εγώ ε, θα, θα ήθελα και δύο. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να πω ότι είναι πρώτη μετά το 2004 είναι η Βόρειος Κορέα της Αφρικής, μια υπαίθρια φυλακή, άνθρωποι που φεύγουν οι νέοι που για να αποφύγουν την επαόριστον ε, στρατιωτική θητεία. Το 2011 αποφάσισε μονομερός να διακόψει τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά σήμερα αποφάσισε να ξανααρχίσει τις σχέσεις. Δεν υπάρχει καμία μοικιό που να μπορεί να εργαστεί εκεί. Πόση βοήθεια θα φτάσει στο πληθυσμό, πώς τα προγράμματα εξηλεκτρισμού μπορούν να εφαρμοστούν χωρίς να ε, ικανοποιούνται συμφέροντα μερικών. Έχει δοθεί υπόσχεση για την στρατιωτική θητεία όταν ε, θέλουμε να εκπαιδεύσουμε τους συνοριοφύλακες ε, μας λένε ότι δεν γίνεται. Αυτό δεν μπορεί να μειώσει την φτώχεια ή να μειώσει το στρες του πληθυσμού όπως και την ένταση στην περιοχή. Είναι το αντίθετο που συμβαίνει. Ευχαριστώ πολύ κυρία Βεργιά. Τώρα εξ ονόματος των Πρασίνων η κυρία Τζούντιθ Σαργεντίνη. Ένα λεπτό κι εσείς. Ευχαριστώ, πολύ. Πρόεδρε. Κάνουμε τη συζήτηση αυτή εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ουδέποτε θεωρώ ότι είχαμε εγκρίνει ομόφωνα ένα πρόγραμμα αναπτυξιακής βοήθειας. Ομόφωνα είχαμε ταχθεί κατά, αλλά από ό,τι φαίνεται το Συμβούλιο δεν το έλαβε υπόψη του καθόλου αυτό. 200 εκατομμύρια ευρώ ήταν το ύψος του προγράμματος αυτού που υποτίθεται ότι θα χρησιμοποιούνται τα ποσά αυτά κατά της παράνομης μετανάστευσης. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί Ερυθρέοι οι οποίοι φεύγουν από τη χώρα τους ακριβώς επειδή λιμοκτονούν. Αν καταφέρουν να επιζήσουν κατά τη διάρκεια του επικίνδυνου αφού ταξιδιού θα πρέπει να καταφέρουν καταρχάς να ξεφύγουν από τους συνοριοφύλακες, πολλοί εκ των οποίων τους, τους πληροβολούν και στη συνέχεια θα πρέπει να καταφέρουν να φτάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάρα πολλές φορές όμως πέφτουν θύματα εκβιασμού και στα πλαίσια του φορολογικού συστήματος όπως είπαμε. Σαφώς λοιπόν χρειαζόμαστε μια συμφωνία με την Τουρκία αλλά πρέπει να είμαστε και πάρα πολύ προσεκτικοί πως διεξάγουμε το διάλογο και την προστασία των συνόρων. Ο κύριος με έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έξι εκατομμύρια περίπου είναι οι κάτοικοι της Ερυθρέας και ξέρετε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί οποίοι προσπαθούν να περάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Μένο Βασίλειο. Και αυτό έχει να κάνει με την στρατιωτική δικτατορία που υπάρχει στην χώρα αυτή που ουσιαστικά επιβάλλει μια στρατιωτική θητεία που ισοδυναμεί με καταδικαστική εργασία. Για ποιο λόγο λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση θεώρησε ότι θα πρέπει οικονομικά να τονώσει αυτούς τους δεσπότες της Ερυθρέας οι οποίοι ουσιαστικά προωθούν μια ολοκληρωτική κυβέρνηση χωρίς καμία λογοδοσία και χωρίς να υπάρχει κράτος δικαίου. Πραγματικά αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι ξοδεύει και σπαταλά τα χρήματα των Βρετανών φορολογούμενων η Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να συνειδητοποιεί τελικά πού βρίσκονται τα βαθύτερα αίτια της κρίσης της χώρας αυτής. Ε, ε, Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρος. κύριος Βέντα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε πρόεδρε. Το 1993 ανέξε την ε, ανεξαρτησία της η Ερυθρέα και αυτό μας έδινε ελπίδες για δημοκρατία. <clears throat> και το Σύνταγμα μετά τόνισε το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ποτέ όμως δεν εφαρμόστηκε, δεν έχουν γίνει ποτέ εκλογές στη χώρα αυτή. Είναι ένα ολοκληρωτικό καθεστώς με κανένα σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα, σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση οικονομικά, με θυγόμενο από πολλές ε, καταστάσεις ξηρασίας και όλα αυτά έχουν οδηγήσει σε μαζική μετανάστευση υπολογίστε ότι κάθε μήνα φεύγουν 5.000 άτομα από τη χώρα αυτή. Το πρόγραμμα ανάπτυξης το οποίο ενεκρίθη είναι μονάχα ένα μικρό βήμα για να μπορέσουν να βοηθηθούν οι πολίτες της χώρας αυτής. Μπορεί να μειώσει την ένδια, αλλά δεν θα λύσει όλα τα προβλήματα που υπάρχουν στη χώρα αυτή. Για να μπορέσει να υπάρξει ανάπτυξη πραγματική στην Ερυθρέα θα πρέπει να γίνουν διαφορετικές αλλαγές στη χώρα αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και ο πρόεδρος κυρία Λίντα Μακέιβαν. Ένα και μισό λεπτό. Κυρία Υπουργέ, ως πρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης είμαι υπερήφανη για μερικά μέτρα ε, για να βεβαίως δεν είναι ένα από τα θέματα αυτά η Ερυθρέα διότι ακούσατε να γίνεται για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είναι φρικτή στην Ερυθρέα. Γι' αυτό τον Νοέμβριο η Επιτροπή μας ομόφωνα ζήτησε να μην ληφθεί απόφαση για νέο πρόγραμμα χωρίς περαιτέρω διάλογο με το Κοινοβούλιο και με τους Υπουργούς. Ε, αλλά ε, προχωρήσατε, υπογράψατε το πρόγραμμα και δεν αγνοήθηκε μόνο η γνώμη ε, της, του Κοινοβουλίου αλλά και της Επιτροπής μου. Δεν είναι καλή αυτή η συμπεριφορά της Κομισιόν. Ελπίζω να μην ξανασύμβει. Πρόκειται για μια σοβαρή απόφαση και ελπίζω ότι όταν ε, το ετήσιο πρόγραμμα δαπανών ε, αποφασιστεί θα εμπλακούμε και εμείς στη συζήτηση. Είπατε ότι θα καταπολεμηθεί η πτώχεια, αλλά 95% χορηγείται για ενεργειακά προγράμματα. Αλλά πού κατευθύνονται τα χρήματα. Δεν υπάρχει ιδιωτικό τομέα στην Ερυθρέα. Πού πηγαίνουν τα χρήματα. Αυτό θέλουμε να μάθουμε σχετικά με την με κρίση των προσφύγων, ο αριθμός των πολιτών της Ερυθρέας στη χώρα μου έχει μειωθεί. Αυτοί που έρχονται ως πρόσφυγες είναι λόγω του πολιτικού συστήματος. Δεν είναι μετανάστες και δεν θα πρέπει να συνδέουμε μεταξύ την, τις σχέσεις μας με την Ερυθρέα με τον αριθμό των προσφύγων που έρχεται από αυτή τη χώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα δίνω τον λόγο. Κυρία Μακέβεν, δέχεστε μια μπλε κάρτα. Δέχεστε μπλε κάρτα, κυρία Μακέβεν. Από τον κύριο Βεστόφσκι. Ναι ή όχι. Ναι. Έχετε την άδεια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ίσως έχετε δίκιο όταν λέτε ότι η βοήθεια στην Ερυθρέα δεν θα ε, κατευθυνθεί στους στόχους και δεν θα υπάρχουν κοινωνικά πλεονεκτήματα από την βοήθεια. Ποιο είναι το πόρισμά σας, έχετε καμία ιδέα θετική για αυτήν την βοήθεια για την Ερυθρέα, πώς να ελέγξουμε τις δαπάνες αυτές, αν τα χρήματα ε, δεν ε, πάνε στους σωστούς στόχους. Δώστε μας μια εναλλακτική λύση αντί να κάνετε κριτική. Ποια είναι η γνώμη σας. Απάντηση. Ευχαριστώ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνομιλήσει κανείς με μια κυβέρνηση που έχει τέτοια φεκτή κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πώς πρόγραμμα βοήθειας με τέτοια κυβέρνηση. Ε, έχουμε συμφωνήσει ένα πλαίσιο. Δεν έχουν χορηγηθεί χρήματα. Προτού χορηγηθούν χρήματα θα πρέπει ε, να υπάρξει περαιτέρω συζήτηση και να συμμετάσχει και το Κοινοβούλιο. Αυτό ζητώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα... Δίνουμε τον λόγο στην κυρία Λόλα Λόλα Ντέντι για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ερυθρέας προβλέπει 250 εκατομμύρια ευρώ για ενεργειακά κυρίως προγράμματα, τα οποία καθόλου ή ελάχιστα θα βοηθήσουν την ανακούφιση της ένδυας και αντίθετα θα ωφελήσουν τις μεγάλες ευρωπαϊκές πολιτικές και τη διαφθορά στην Ερυθρέα η Ευρωπαϊκή Ένωση <coughs> έχει υπογράψει τη λεγόμενη Συμφωνία Χαρτούμ για τις χώρες της περιοχής ώστε η Ερυθρέα να είναι μία από τις χώρες η οποία θα είναι σημείο ελέγχου για τις μεταναστευτικές ροές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά είναι μια δικτατορία η Ερυθρέα που παραβιάζει συστηματικά τα ανθρώπινα δικαιώματα και καταστέλει τον πλουτισμό της. Σύμφωνα με την ε, αρμόδια υπηρεσία του ΟΗΕ, το 20% των ατόμων που διασύζουν τη Μεσόγειο προέρχεται από την Ερυθρέα γιατί προσπαθούν να φύγουν από αυτή τη φυλακή. Όλα αυτά τα οποία γίνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά νομιμοποιούν μια δικτατορία για να εξυπηρετήσουν τα γεωστρατηγικά μα συμφέροντα. Και συγχρόνω κλείνουμε τα μάτια στη δραματική κατάσταση που ζει ο πληθυσμό τη Ερυθρέα. Α είμαστε συνεπείς, ας σταματήσουμε να χρηματοδοτούμε τυρανικέ κυβέρνηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Φάμπιο Μάσιμο Καστάλντο. Για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο διάλογο στα πλαίσια τη εξωτερική πολιτική είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό να διαλέγουμε και ποιον συνομιλούμε όμω. Μέχρι στιγμής δεν είναι αξιόπιστη η στάση που κρατά η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στην κυβέρνηση αυτή, η οποία ουσιαστικά έχει υποστηρίξει ακόμα και το Al-Shabaab στη Σομαλία. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι, ανήλικοι πάρα πολλές φορές, οι οποίοι αναγκάζονται να φύγουν από τη χώρα αυτή και οι οποίοι πάρα πολλέ φορέ κρατούνται παράνομα από τη χώρα αυτή με κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για να μην μιλήσω για βασανισμού πολιτικών κρατουμένων ή για εκτελέσει ε, με συνοπτικέ διαδικασίε χωρί να έχει προηγηθεί καμία δίκη. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να δούμε ποια θα είναι η αναπτυξιακή βοήθεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η βασική προπόθεση θα πρέπει να είναι να σημειωθεί κάποια πρόοδο από τη χώρα αυτή. Δεν έχουμε δει μέχρι στιγμή κάτι τέτοιο. Α βοηθήσουμε πραγματικά να μειωθεί η ένδυα στη χώρα αυτή, προκειμένου να μειωθεί και η μετανάστευση. Αλλά χρειαζόμαστε πραγματικά επιτεύγματα από την κυβέρνηση αυτή. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να βοηθηθεί ο λαό τη Ερυθρέα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νομίζω ότι θα πρέπει να έχει μια ξεκάθαρη γραμμή και το έχει πει και στο παρελθόν. Θέλει να βοηθήσει το λαό της Ερυθρέα και θα πρέπει να το λάβει υπόψη στο αυτό το Συμβούλιο. Ε, Κύριος Μωρίς Πόγκα, για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η κατάσταση στην Ερυθρέα είναι ιδιαίτερα κρίσιμη. Κάθε μήνα χιλιάδες Ερυθρέοι φεύγουν από την Ερυθρέα εξαιτία της κατάφορης παραβίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων η ερευνητική έκθεση των Ηνωμένων Εθνών για το ζήτημα αυτό, καθώς επίσης και οι δηλώσεις του ειδικού εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ερυθρέα, καταδεικνύουν πραγματικά ότι έτσι έχουν τα πράγματα. Τα μέλη της Επιτροπής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είπαν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο ότι πραγματικά είναι πάρα πολλές οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα αυτή. Στα πλαίσια του δημοκρατικού ελέγχου που υποτίθεται ότι πρέπει να λαμβάνει η χώρα στα πλαίσια της παροχής αναπτυξιακής βοήθειας για τις χώρες που εντάσσονται στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Αγνοήθηκε όμως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θεωρώ ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν θεμελιώδη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δεν μπορούμε να κάνουμε εκχωρήσεις προς αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να γίνει ένας, έλεγχο όσον αφορά τι παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να σταματήσουν αυτέ τι παραβιάσει. Ευχαριστώ. Και εμεί σα ευχαριστούμε. Μπορείτε να δεχθείτε μία μπλε κάρτα από τον κύριο Σόνι. Δέχεστε μπλε κάρτα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητέ συνάδελφοι, αναφερθήκατε στα ανθρώπινα δικαιώματα και είπατε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να προασπίζουμε αυτά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πάρα πολύ όμως αναφέρθηκαν και στη διαφθορά. Το γεγονός δηλαδή ότι το καθεστώς της Ερυθρέας εκμεταλλεύεται οποιαδήποτε βοήθεια της δίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς όμως να διοχετεύεται συνέχεια βοήθεια αυτή προς τους κατοίκους της χώρας. Ισχύει κάτι τέτοιο και πώς σχετίζεται αυτό με την καταστολή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Νομίζω ότι θα πρέπει περισσότερο να αφαιρθούμε και στο ζήτημα της αιρεσιμότητας. Πέρα από τα ανθρώπινα δικαιώματα να θέσουμε και άλλες προϋποθέσεις όπως η καταπολέμηση της διαφθοράς και ούτε καθεξής. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι εναπόκειται στην κυβέρνηση της Ερυθρέας να αρχίσει να καταπολεμά την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να τηρεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και εμεί θα πρέπει να θέτουμε προποθέσει και απαιτήσει σε σχέση με την αναπτυξιακή βοήθεια που δίνουμε προ την Ερυθρέα. Ευχαριστώ. Και εμεί ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα ο κύριος Ενρίκε Γκερέρο Σαλόμ έχει το λόγο. μισή λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Υπουργέ, Σήμερα το πρωί κάναμε μια μακρά συζήτηση σε αυτό το κοινοβούλιο για την κρίση μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αληθεύει το γεγονός ότι η Ερυθρέα δεν είναι η κύρια αιστεία για τους ε, πρόσφυγες. Έχουμε τη Συρία, έχουμε το Ιράκ, έχουμε άλλες χώρες της περιοχής, αλλά δεν είναι μικρή η συμβολή της Ερυθρέας. Με περίπου 400.000 <clears throat> μετανάστες που είναι το 9% του πληθυσμού της και με 5.000 που βγαίνουν κάθε μέρα από την Ερυθρέα. Όλοι αυτοί συμβάλλουν στο να είναι ο αριθμός των προσφύγων σε όλο τον κόσμο 60 εκατομμύρια. Είναι ισοδύναμο λοιπόν ισοδήμονο αριθμό με τον πληθυσμό του Ηνωμένου Βασιλείου τη Γαλλία. Η περίπτωση Ερυθρέα είναι μια σαφή περίπτωση μια κυβέρνηση που παραδιάζει τι θεμελιώδει ελευθερίε, <clears throat> που διώκει του πολίτε τη, που διώκει τι μη κυβερνητικέ οργανώσει, που καταπατά και αποκλείει οποιαδήποτε χρήση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και που δεν εφαρμόζει τους, ε, την απαγόρευση των βασανισμών. Πρέπει να είναι κριτική η στάση μας, αλλά θα πρέπει αυτή η κριτική να συνδέεται και με τη βοήθειά μας. Δηλαδή η βοήθειά μας θα πρέπει να εξαρτάται από το ότι η Ερυθρέα θα δεσμευτεί να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα προβλήματα. Αλλιώ επαναλαμβάνω αυτά που είπε η πρόεδρος της Επιτροπής μας, το Κοινοβούλιο δεν πρέπει να παραγνωρίζεται <clears throat> στη διαδικασία ανάπτυξης έναντι της ΕΕ αλλά πρέπει να είναι ενεργό τμήμα αυτής της προσπάθειας. Ευχαριστώ. Ακολουθεί η κυρία Μαρία Γκαβριέλ. Να Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ. Η κατάσταση στην Ερυθρέα δείχνει πολύ καλά το διακύβευμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση την συνεκτικότητα της αναπτυξιακής πολιτικής με τα ανθρώπινα δικαιώματα και το προσφυγικό και πώς ε, τα μέσα μας θα πρέπει να είναι μέσα πίεσης και μοχλός για να ε, ούτως ώστε να εκδημοκρατιστεί αυτή η χώρα δύο παρατηρήσεις. Ας χρησιμοποιήσουμε καλύτερα ε, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Το Κοινοβούλιο έχει κάνει έκκληση ούτως ώστε το εθνικό πρόγραμμα, κυρίως το φάκελος διακυβέρνησης, να βασίζεται στις αρχές εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης και ούτως ώστε η Ερθρέα να γίνει πιο σταθερή και πιο ανοιχτή μέσα στα πλαίσια του προσφυγικού. Η Ερυθρέη το 2014 ήταν η δεύτερη ομάδα ατόμων που έφτασαν μετά τους Σύρους στην Ιταλία το Ταμείο, ε, η διαδικασία του Χαρτούμα και η Συμφωνία του Κοτονού θα πρέπει να ενεργοποιηθούν για λύσεις κυρίως υπέρ των Ερτρέων πολιτών και των βασικών τους δικαιωμάτων. Βεβαίως, οι αιτίε ε, του, του προσφυγικού είναι σε εκείνη χώρα. Η Ερτρέα είναι ένα παράδειγμα που μπορούμε να κινητοποιηθούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να να καλωσορίσω την αντιπροσωπή από τη Σολινταρνόσκ που βρίσκεται στο θεωρείο. Σας καλωσορίζω όλους. Και τώρα δίνω τον λόγο στην κυρία Άννα Γκόμες. μισή λεπτό. Οι συστηματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ερυθρέα <clears throat> που οξύνονται με την πρακτική της μόνιμης στρατιωτικής θητείας που οδηγεί σε ένα καθεστώς δουλείας, οδηγεί σε 5.000 Ερυθρέ, πολίτες Ερυθρέας που πηγαίνουν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε μήνα φτάνοντας στο συνολικό αριθμό των 400.000 προσφύγων. Δεν υπάρχει καμία έννοια δικαίου, δεν υπάρχει δικαιοσία που λειτουργεί, δεν υπάρχει ανεξάρτητη, ε, ανεξάρτητος τύπος και μεσανημένως δεν υπάρχουν μη κυβερνητικές οργανώσεις. Και παρόλα αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να δώσει βοήθεια 250 εκατομμυρίων σε μια δικτατορία για να πετύχει, να σταματήσει το, τη μεταναστευτική ροή. Μα πώς μπορεί η Κομισιόν να φαντάζεται ότι ένα τέτοιο σχέδιο μπορεί να βοηθήσει να βελτιώσει συνθήκες διαβίωσης του πληθυσμού στην Ερυθρέα αυτή η βοήθεια λοιπόν μέσα στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης και παρά την αντίθετη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όλα αυτά δείχνουν ότι δεν υπάρχει δημοκρατικός έλεγχος σε αυτό το Ταμείο και δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί για κανένα άλλο στόχο όπως η αγορά όπλων, η αποσταθεροποίηση της περιοχής και η περαιτέρω καταπίεση του λαού της Ερυθρέας. Θα πρέπει η Κομισιόν να δρά σε ένα ελάχιστο επίπεδο σε ό,τι αφορά τη δημοκρατία και να εξασφαλίζει ότι τα σχέδια που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ελέγχονται από ανεξάρτητους οργανισμούς και υπάρχει πρόσβαση μη κυβερνητικών οργανώσεων και του ειδικού εισηγητή των Ηνωμένων Ευχαριστώ κυρία Βουλευτά. Ο κύριος Ιωακίμ Τσέλερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι φεύγουν από την Ερυθρέα γιατί υπάρχει εκεί μια δικτατορία η οποία φτάνει μέχρι την τελευταία γωνιά της καθημερινής ζωής. Η Κομισιόν παρόλα αυτά έδωσε 200 εκατομμύρια ευρώ για ένα εθνικό ενδεικτικό πρόγραμμα και από τα οποία 20 εκατομμύρια για ευκυβερνησία. Αυτό αν είναι αστείο. Ήδη εδώ και καιρό το 10ο Αναπτυξιακό Ταμείο έδωσε 200 εκατομμύρια στην ε, Ερυθρέα, αλλά μειώθηκαν τα ποσά αυτά σε 35 εκατομμύρια γιατί δεν υπήρξε καμία απολύτως πρόοδος για τα θέματα αυτά. Το 2014 πήγε μια ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία στον Ερυθρέα και είπε ότι κανένα από τα προγράμματα αυτά δεν λειτουργούσε, επομένω τα χρήματα αυτά δεν πρέπει να δοθούν και δεν πρέπει η Κομισιόν να δώσει καθόλου πρόσθετα ποσά προ την Ερυθρέα. Εδώ έχουμε μια περίπτωση όπου το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη θα πρέπει επιτέλου να τεθεί κάτω από κοινοβουλευτικό έλεγχο και η γνωμοδότησή μας κινείται ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ, λέει και ο πρόεδρος. Η κυρία Μαρίτα Ουλσκοκ. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε, κυρία Υπουργέ. 5.281 μέρες. Κρατάτε ο Νταβίτ Ισάκ, ο Ερυθρέος δημοσιογράφος, 5.281 ημέρες. Πάνω από 14 χρόνια αβεβαιότητας, απόγνωσης, άγχους για την οικογένειά του. Είναι ο μόνος Ευρωπαίος υπήκος, ο οποίος είναι φυλακισμένος για τις απόψεις του αυτή τη στιγμή και Βέβαια, υπάρχουν και πολλοί άλλοι πολιτικοί κρατούμενοι στη χώρα αυτή που αντιμετωπίζουν προβλήματα, γιατί ξέρετε ότι η κυβέρνηση βάλει κατά τη ε, ελεύθερη έκφραση και το έχει πει αυτό και ο ειδικό απεσταλμένο των ΗΕ, ο ειδικό συγητή των ΗΕ. Συνεχεί και συστηματικέ παραβιέ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ξέρετε ότι έχει περιορίσει πάρα πολύ τι ελευθερίε των πολιτών η κυβέρνηση αυτή. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Όσον αφορά λοιπόν τη δική μα τώρα την εξωτερική πολιτική, θέλουμε να προωθήσουμε το κράτο δικαίου, να προωθήσουμε τη δημοκρατία, βασικέ και θεμελιώδει θεμελιώδει ελευθερίε, πολύ ωραία. Αυτή είναι η βασική μα αποστολή, αλλά θα πρέπει αυτό να ισχύει και για τη σχέση που έχουμε με την Ερυθρέα. Είμαι υπέρ του ψηφίσματο, αλλά θα ήθελα να ξέρω ακριβώ ποια είναι η άποψη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι ακριβώ πρέπει να κάνετε για την περίπτωση του Νταβίτη Σάκ, του δημοσιογράφου αυτού. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα το λόγο έχει για ένα λεπτό ο κύριο Λάρ Αντάκτουσον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Υπουργέ να σας ευχαριστήσω πραγματικά για αυτή την πάρα πολύ καλή σύνοψη και παρουσίαση που μας κάνατε για την Ερυθρέα και να σας ευχαριστήσω για την υποστήριξη που μου δώσετε σε σχέση με τον Νταβίτ Ιζακ, τον Σουηδοερυθρέο δημοσιογράφο, ο οποίος για πάνω από 14 χρόνια βρίσκεται σε φυλακές της Ερυθρέας σε απάνθρωπες συνθήκες. Και ο μόνος λόγος για τον οποίο ο άνθρωπος αυτός είναι φυλακισμένος είναι το ότι υπερασπίστηκε τα ανθρώπινα δικαιώματα το ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά τώρα την άμεση απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Παράλληλα όμω πρέπει να γίνουν περισσότερα πράγματα. Οι παραβιάσει αυτέ ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αν συνεχιστούν ανεμπόδιστε, αυτό προφανώ θα έχει πολύ σημαντικέ επιπτώσει για την ε, διεθνή συνεργασία που θέλουν να έχουμε με τη χώρα αυτή. Δεν είναι ποτέ δυνατό η Ευρωπαϊκή Ένωση να δίνει στην Ερυθρέα χρήματα χωρί προποθέσει. Πρέπει να έχουμε ρεσιμότητα, πρέπει να έχουμε προποθέσει. Και μία από τι προποθέσει αυτέ είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα και η απελευθέρωση του Ταβίτη ΣΑΚ. Και βέβαια και οι υπόλοιποι πολιτικοί κρατούμενοι θα πρέπει να απελευθερωθούν. Α μην ξεχνάμε και ας μην παραβλέπουμε ότι η Ερυθρέα δυστυχώς είναι ένα διεφθαρμένο κράτος. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Ντόρου Κλαούντιαν Φουντσούλιτσα. Για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μιλάτε κυρίες και κύριοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να ξαναδώσει βοήθεια στην Ερυθρέα με ένα ενδεικτικό πρόγραμμα που αναφέρεται σε 200 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά αυτό την ίδια τη στιγμή που η ομάδα Α της Επιτροπής ε, της ζήτησε το Νοέμβριο του 2015 η Επιτροπή της οποίας προεδρεύω το σχέδιο αυτό να μην υιοθετηθεί ε, αμέσως. Ε, αλλά βεβαίως η γνώμη του Κοινοβουλίου δεν έχει καμία σημασία, δεν λαμβάνεται υπόψη. γιατί έχουμε δώσει μια γνώμη αρνητική λόγω της συνεχούς επιδείνωσης της εσωτερικής κατάστασης στην Ερυθρέα. Υπάρχουν συνεχώς αυθαίρετες συλλήψεις. Οποιοςδήποτε κατακρίνει την κυβέρνηση συλλαμβάνεται, οποιοςδήποτε θέλει να κάνει το δημοσιογράφο ε, φυλακίζεται λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες στρατολόγησης, οι στρατολογημένοι ε, φεύγουν ε, μαζικά και οι Ερυθρέοι είναι η τρίτη μεγαλύτερη ομάδα που φτάνει στην Ευρώπη. Πρέπει οι αποφάσεις μας να λαμβάνονται υπόψη από το Συμβούλιο και από την Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Τώρα έχουμε την διαδικασία ε, Catch the Eye, ο κύριος Μπραν Χάιες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ελπίζω να επισκεφθώ την Ερυθρέα τις επόμενες εβδομάδες με μια ΜΚΟ Β την Ιρλανδική που ασχολείται με την ανάπτυξη και ελπίζω να μεταδώσω το μήνυμα του ψηφίσματος που θα περάσει ελπίζουμε αύριο. Πρέπει να εξασφαλίσουμε την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να καταπολεμηθεί η διαφθορά στην Ερυθρέα και ε, να δούμε ότι ε, η χρηματοδότηση στην Ερυθρέα πρέπει να πηγαίνει στον πληθυσμό της Ερυθρέας για να ωφεληθεί ο πληθυσμός και κανείς άλλος. Και νομίζω ότι ένα δυνατό μήνυμα σε εσά κυρία Υπουργέ, στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο, είναι ότι πρέπει να υπάρχει αιρεσιμότητα ε, και η χρηματοδότηση που θα δώσουμε στην Ερυθρέα και σε άλλα μέρη του αναπτυσσόμενου ε, κόσμου να βασίζονται στα ανθρώπινα δικαιώματα, ούτω ώστε η κυβέρνηση να δεχθεί να fide. Ε, συμφωνώ με όσους είπαν είναι ότι για την πρόταση την περιεκτική αλλά θα πρέπει να μιλήσουμε για την ανάγκη να υπάρξει πρόεδρος όσον αφορά την απελευθέρωση του Νταβίντ Ισάκα και θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι η χρηματοδότηση προς την Ερυθρέα θα πρέπει να ωφελεί τον πληθυσμό της Ερυθρέας και κανέναν άλλο. Ο κύριος Νικόλα Καπούτο τώρα το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Ερυθρέα είναι χώρα προέλευσης πάρα πολλών προσφύγων που φτάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με το Human Rights Watch, η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι τεράστια. Εκτελέσεις χωρίς να γίνονται δίκες, βασανιστήρια, καταναγκαστική εργασία. Από έκθεση των ΗΕ βλέπουμε ότι η α, κυβέρνηση αυτή συνεργάζεται πολλές φορές ακόμα και με γειτονικέ χώρες προκειμένου να προχωρήσει στην παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι συνθήκε είναι τόσο άθλιε στην χώρα που η Amnesty International ζήτησε από πάρα πολλέ χώρε να σταματήσουν οποιαδήποτε συνεργασία που έχουν με τη χώρα αυτή. Και μάλιστα αυτό απασχόλησε και την σύνοδο τη Ευρωπαϊκή Ένωση με την Τουρκία όσον αφορά τη διαχείριση των προσφυγικών ροών που έρχονται και από τη χώρα αυτή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να βελτιώσουμε τι θεμελιώδει ελευθερίε στη χώρα αυτή προτού προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε άλλη συνεργασία. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε και εμεί πολύ. Ο κύριος Μαριάς τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σύμφωνα με το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, στην Ερυθρέα παρατηρούνται συστηματικές και σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Ερυθρέα έχει να διεξάγει δημοκρατικές εκλογές από το 1993. Από το 2001 υπάρχει στη χώρα καθεστώς δικτατορίας, ενώ παράλληλα το 5% του πληθυσμού έχει εγκαταλείψει τη χώρα λόγω πολιτικής κατάστασης και οικονομικής δυσχέρειας επιπλέον στην ερυθρέα παρατηρούνται περιορισμοί στην ελευθερία λόγου και ελευθεροτυπίας καθώς και στην θρησκευτική ελευθερία ενώ κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας σημειώνονται συχνά βασανιστήρια και εκτελέσεις. απέναντι στην παραβίαση δικαιωμάτων που λαμβάνει η χώρα στην ερυθρέα θα πρέπει η ευρωπαϊκή ένωση να συμβάλει στην προώθηση ενός δημοκρατικού μοντέλου διακυβέρνησης. παράλληλα κάθε κράτο μέλο της ένωσης οφείλει να καταδικάσει την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και τη σύνδεση μεταξύ επιχειρήσεων κυβέρνηση και διαφθοράς τέλος η ευρωπαϊκή ένωση θα πρέπει να αναθεωρήσει την επενδυτική πολιτική της στη χώρα και να συμβάλει στην καταπολέμηση των ανισοτήτων και της φτώχειας στην περιοχή. ευχαριστώ. ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. εδώ και πολλά χρόνια τώρα πια έχουμε παρακολουθήσει τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ερυθρέα. Διάφορες μορφές δουλείας του πληθυσμού εκεί. Έλλειψη της ελευθερίας άσκησης θρησκευτική συνείδησης. Βία κατά των γυναικών. Απόλυτη <clears throat> απουσία σεβασμού για την κοινότητα των ΛΟΑΔΜ η φυλάκιση πολιτών ακόμα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολλές άλλες περιπτώσεις που στοιχειοθετούν την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρέπει να βοηθήσουμε την Ερυθρέα. Ναι, πρέπει να τη βοηθήσουμε, αλλά τονίζουμε όλοι μας ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει το λαό τη Ερυθρέα. Το θέμα είναι αν είμαστε πράγματι σε θέση να το κάνουμε αυτό. Μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα χρήματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν προ αυτό το σκοπό <clears throat> και δεν θα χρησιμοποιηθούν προ όφελος του δικτατορικού καθεστώτος. Ο κύριος Κάρβερ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ερυθρέα είναι μια χώρα που αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις πολιτική αστάθεια, παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δια της βίας στρατιωτική θητεία. Όλα αυτά έχουν οδηγήσει στην ανθρωπιστική κρίση που γνωρίζουμε. Είναι από τις κύριες πηγές μεταναστών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλές χιλιάδες κάνουν αυτό το επιχείρημα ταξίδι για να πάνε στην Ευρώπη. Με την Αιθιοπία και το Σουδάν και την Ιεμένη στα σύνορά της, δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε το ρόλο της Ερυθρέας. Πάνω από 35.000 Ερυθρέοι ε, πρόσφυγες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Αιθιοπία και παίζει σημαντικό ρόλο η Αιθιοπία στον αγώνα κατά της Al-Shabaab. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα λοιπόν για να αντιμετωπίσουμε τους λόγους που οδηγούν στην ροή των προσφύγων από την Ερυθρέα. Και μόνο με στενή συνεργασία με περιφερειακές δυνάμεις μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα με αποτελεσματικό και γρήγορο τρόπο. Και για το λαό της ε, μέσα Ανατολής και για το λαό του κέρατος της Αφρικής και το λαό της Ευρώπης. Uh, thank you um, now, uh... Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, εξ ονόματος της ε, κυρίας Μογκερίνη, το λόγο έχει η Υπουργός Ζανίν Χένις Πλασέρτ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως σας είπα ήδη στην αρχική μου παρέμβαση, μας προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία η ε, συνεχόμενη, συνεχιζόμενη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα αυτή. Αντιμετωπίζουμε λοιπόν σε όλου τι συναντήσει που έχουμε με τους υπουργού το ζήτημα αυτό τη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σε επαφή με την κυβέρνηση αυτή και στα πλαίσια διεθνών φόρα και ιδίω στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με το Εθνικό Ενδεικτικό Πρόγραμμα το οποίο εγκρίθηκε, θα γινόντουσαν απαραίτητε τροποποίησει στη στάση την οποία κρατάει η Ερυθρέα όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα μπορούσαμε να βαθύνουμε περισσότερο το διάλογο που έχουμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα με την κυβέρνηση αυτή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσβλέπει λοιπόν σε μια εταιρική σχέση με την Ερυθρέα προκειμένου να γίνουν περισσότερε παραχωρήσει και από τι δύο πλευρέ. Αυτό είναι η αιρεσιμότητα. Γι' αυτό ακριβώ το λόγο έχουμε πει στην κυβέρνηση Ερυθρέα ότι θα πρέπει η συνεργασία μα να συνοδεύεται από από συγκεκριμένες δράσεις και συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να έχουν να κάνουν με την εφαρμογή των συστάσεων που έχουμε κάνει. Να βελτιωθεί η δημόσια διοίκηση και η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Από το 2016 μέχρι το 2020 θα γίνουν επεμβάσεις σε διάφορους τομείς όπως ο τομέας της ενέργειας και αυτό θα αποτελέσει προϋπόθεση προκειμένου να προστατευτεί περισσότερο η γεωργική παραγωγή και να προωθηθεί η επισητιστική ασφάλεια. Θέλουμε να δημιουργήσουμε επίσης καλύτερες συνθήκες για μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Επιθυμούμε μέσω της συνεργασίας αυτής να προστατεύσουμε και την ευημερία των ε, Ερυθρέων και να μειώσουμε τα φαινόμενα φτώχειας. Επιθυμούμε επίση να βελτιώσουμε προφανώ τα ανθρώπινα δικαιώματα στα πλαίσια του προγράμματο αυτού και γι' αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να υποστηρίζει τι συστάσει που έχουν γίνει προ την Ερυθρέα στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών και τη περιοδική αναθεώρηση των Ηνωμένων Εθνών. Τώρα, όσον αφορά το ζήτημα της αναπτυξιακής βοήθειας και άκουσα πάρα πολλές σχετικές παρατηρήσεις. Η αναπτυξιακή βοήθεια δίδεται βάσει συγκεκριμένων σχεδίων που έχουν ως στόχο να βοηθήσουν και την κατάσταση των ανθρώπων στην Ερυθρέα, να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης, να μειώσουμε την ένδια. Δεν υπάρχει καμία υποστήριξη προς την κεντρική κυβέρνηση. Θέλουμε να προωθήσουμε τα ευρωπαϊκά αυτά προγράμματα με τρόπο απόλυτα διαφανή, ακολουθώντας τους κανόνες που διέπουν τόσο τα ευρωπαϊκά προγράμματα ανάπτυξης όσο και τα προγράμματα ανάπτυξης των μένων εθνών και υπάρχει μια συνεχής παρακολούθηση και εποπτεία των προγραμμάτων αυτών από τις αρμόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δικαιούχοι της χρηματοδότησης αυτής είναι οι ίδιοι Ερυθρέοι. Το τονίζω για μία ακόμη φορά. Σε καμία περίπτωση δεν υποστηρίζουμε την κεντρική κυβέρνηση της χώρας. Κύριε Πρόεδρε, Γνωρίζω πάρα πολύ καλά, όπω το είπαν και πάρα πολλοί συναδελφοί σα, ότι όντω το πολιτικό καθεστώ είναι πάρα πολύ δύσκολο στη Ερυθρέα και το πολιτικό πλαίσιο στο οποίο δραστηριοποιούμε θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θέλουμε λοιπόν ανατακτά χρονικά διαστήματα να ερχόμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πραγματικά να κάνουμε ένα απολογισμό του κατά πόσο σημειώνει πρόοδο η κυβέρνηση αυτή στις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να κάνει. Η κυρία Μογκερίνη δεσμεύεται λοιπόν αντακτά χρονικά διαστήματα να ενημερώνει αναλόγω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σα διαβεβαιώ ότι θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυ στην εξέλιξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ερυθρέα και το ρόλο που διδραματίζει η χώρα αυτή στην ευρύτερη περιοχή. Όπω είπα στην αρχική μου παρέμβαση, δεσμευόμαστε με την Ερυθρέα, συνεργαζόμαστε με την Ερυθρέα για να βοηθήσουμε του ανθρώπου. Περαιτέρω απομόνωση τη χώρα αυτή σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να βοηθήσει του Ερυθρέου. Σα ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Υπουργέ. Έχω λάβει 7 ψηφίσματα, προτάσεις ψηφίσματος από όλες τις πολιτικές ομάδες ουσιαστικά και για το κλείσιμο της συζήτησης η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο.